Συγγνώμη, ξέχασα να ανάψω το μικρόφωνο μου. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Νινέτ Κέλλη, εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες στον Λίβανο. Θα μας μιλήσει για την κατάσταση των σύρων προσφύγων στο Λίβανο. Επαναλαμβάνω, η κυρία Κέλλη εκπροσωπεί στο Λίβανο την της αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Είναι εκατομμύρια οι Σύριοι πρόσφυγες που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο από τη Συρία. Υπολογίζονται στα 4 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από τη Συρία. Τεράστια η ανησυχία που προκαλεί η ανθρωπιστική κατάστασή τους και κυρίως ε, τα 2 εκατομμύρια νέων ανηλίκων για την ακρίβεια, <coughs> κάτω των 18 ετών. Είναι μια ολόκληρη γενιά που μπορεί να πάει στράφη. Επίσης, 100.000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια έχουν γεννηθεί στην εξορία και με βάση την ε, νομοθεσία της Συρίας ε, μπορεί να χαρακτηριστούν απάτριδες. Η κυρία Κέλλη θα μας κάνει μια παρουσίαση της κατάστασης των προσφύγων ε, στο Λίβανο αυτή τη στιγμή θα ήθελα να τη συγχαρώ και για το δικό της έργο, αλλά και για το έργο της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια, η κυρία Λόχ Μπιλερ και ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ που μόλις επέστρεψαν από την περιοχή, θα μας κάνουν τη δική τους ενημέρωση. Κυρία Κέλλη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, ανάμεσά σας, για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, όταν κανεί δουλεύει στον Λίβανο και αντιμετωπίζει αυτού του είδους ε, τις ανθρώπινες απίστευτες τραγωδίες ε, μετά από τέσσερα χρόνια στη Μέση Ανατολή κανείς ξεχνάει πως είναι υπόλοιπος κόσμος επομένως με ευχαριστεί πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και βέβαια θα πρέπει να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ όσον αφορά τις ε, ανθρωπιστικές προσπάθειες ό,τι έχει γίνει στον ε, Λίβανο. Τώρα όπως είπαμε ξεκινάει η τέταρτη χρονιά μας εκεί και ό,τι και να πω είναι λίγο για το πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά. Ε, να είστε βέβαιοι, σας ευχαριστεί και ο κόσμος όλη την ώρα και ε, δεν λέω τίποτα παράξενο αλλά αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ότι από νωρίς κατά την κρίση ήταν την ανάγκη, τη διέβλωση ανάγκη, η ανθρωπιστική ανάγκη υποστήριξη, βοήθεια, ούτως ώστε εμείς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανάγκες των προσφύγων. Αλλά πιο σημαντικό να μπορέσει ο Λίβανος να ανταποκριθεί σε αυτή την τρομερή τραγωδία. Σήμερα να σας εξηγήσω τι γίνεται εκεί, ποια είναι τα βασικά θέματα, τα βασικά προβλήματα. Αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η σταθερότητα της χώρας. Μιλούμε για πάνω από ένα εκατομμύριο προσφύγων που ήρθαν και τα πράγματα σε μια έφραυστη ισορροπία. Άρα πάρα πολύ σημαντική υπόθεση η ελληνική και επομένως βλέπετε αυτό την πρώτη διαφάνεια τι έγινε εδώ από το 2011 είχαμε 2.000 πρόσφυγες στον Ιούνιο τότε η, η χώρα ε, αριθμεί 4 εκατομμύρια κατοίκους ε, και όσοι έχουν επισκεφτεί τη χώρα ε, έχουν καταλάβει πόσο μικρή είναι και σε ένα χρόνο ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε από 25.000 σε... Α, μισό λεπτό, πάμε στο επόμενο. Από 2.000 λέει ο Μιλήτρη. από 2.000 πήγε στις 25.000. Αλλά μεταξύ 2012 και 2013 έγινε το άλμα. Είχαμε μισό εκατομμύριο προσφύγων στον Λίβανο. Ε, φυσικά αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλοι αυτοί κατέκλυσαν τη χώρα και συνεχίστηκε αυτή η τάση και φτάσαμε στο 1 εκατομμύριο και παραπάνω τον Ιούνιο του 2014. Σήμερα τι γίνεται. Έχουμε 1.183.000 πρόσφυγες και αν προσέξετε λίγο αυτόν τον χάρτη θα διακρίνετε ότι έχουμε κάποιες ε, περιοχές που είναι λευκού χρώματος. Αυτά είναι τα βουνά στο κέντρο. Και επίσης προς Ανατολάς, εκεί που είναι κάποιες ε, περιοχές ε, διαφλενικούμενες και μπορείτε να δείτε ε, την τάση σε αυτό το γράφημα ότι έχουμε κάπως πτωτική τάση γιατί άρχισε από την κυβέρνηση ε, κάποια περιοριστική πολιτική να μην μπαίνουν τόσο πολύ στη χώρα. Για κοιτάξτε τώρα εδώ για να καταλάβετε καλύτερα. Κοιτάξτε. Το Λίβανο σε σχέση με το μέγεθος του Βελγίου. Για να καταλάβετε πώς είναι για μια μικρή χώρα σε 18 μήνες πάνω από ένα εκατομμύριο συν πρόσφυγες. Πάνω από ένα εκατομμύριο δηλαδή. Οπότε Να μην επίσης ξεχνούμε και το ποσοστό, δηλαδή μιλούμε για το 1 τέταρτο του πληθυσμού και παραπάνω. Γιατί έχουμε επίσης 280.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα. Εδώ και χώρα και έχουμε και 43.000 Σύρους πρόσφυγες. Παλαιστίνιους της Συρίας. Βλέπετε εμάς ότι πρόκειται για μαζική, για τεράστια μετακίνηση πληθυσμού προς τον Λίβανο που έχει επομένως πάρα πολύ σοβαρές ε, οικονομικές συνέπειες υποστεί γιατί υπήρχαν εμπορικές ζωές πολύ σημαντικές με τη Συρία ε, οπότε χτυπήθηκε το εμπόριο, χτυπήθηκε η κατανάλωση, πέσανε οι επενδύσεις και όλα αυτά ήταν πολύ κακά για την οικονομία. Και πέραν τούτου έχουμε την άφηξη των προσφύγων. Ένα εκατομμύριο είπαμε οι οποίοι επίση έφεραν σε πολύ δύσκολη χώρα, στρίμωξαν αυτή τη χώρα η οποία ήδη είχε προβλήματα με την διοίκηση και τι κρατικέ υπηρεσίε. Για κοιτάξτε τώρα, το θέμα ποια είναι η κρατική πολιτική. Εδώ είναι το τι συμβαίνει. Δεν έχετε δει στι ειδήσει τίποτε διαμαρτυρίε, αντιπαραθέσεις, διαδηλώσει κατά των προσφύγων. Αυτό ε, λέει ακριβώς το πώς ανταποκρίθηκαν, πώς αντέδρασαν οι Λιβανέζοι αυτή την κρίση. Τόση γενεδορία δεν έχω δει στη ζωή μου πουθενά. Ακόμα και τώρα που έχουμε κάποιες εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, παρόλα αυτά υπάρχει συγκράτηση και αυτοσυγκράτηση. σε κάποιες κοινότητες, σε κάποιες ε, δήμους και κοινότητες, έχει πιο πολλούς πρόσφυγες από τους κατοίκους και λέει, τους αντιμετωπίζουν ως αδελφούς και αδελφές και λένε πρέπει να τους προστατεύσουν. υπήρξαν πολιτικά προβλήματα τότε που άρχισε η κρίση. Α βλέπετε και σε αυτό το διάγραμμα ότι είχα μια υπηρεσία για κυβέρνηση σε κάποιες φάσεις όπου υπήρχε κάθετη αύξηση των προσφύγων. Αυτό σημαίνει ότι τότε δεν ήταν δυνατόν ούτε να θεσπιστούν νόμοι ούτε να ασκηθεί κάποια ουσιαστική πολιτική. Μάιο 2014. Βλέπετε τότε έληξε η θητεία του Προέδρου. Έχει κυβέρνηση αλλά μόνο συνετικά μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Επομένως βλέπουμε ότι πάλι εμποδίζεται η χάραξη πολιτικής μια που υπάρχει τόση αστάθεια. Επίσης, τον Οκτώβριο κατάφεραν να συγκεντρώσουν κάποια συνένεση για ενιαία πολιτική, για πολιτική. Βλέπουμε, να αυτή είναι η πολιτική. Μία σελίδα με τέσσερι, τέσσερις αρχές. Πρώτα από τα μία συμφωνία ότι η κυβέρνηση και η χώρα δεν μπορούν να υποδεχθούν άλλους πρόσφυγες. Μια που έχουν φτάσει στο 25% του πληθυσμού. Δεύτερον, για κοιτάξτε την άλλη διαφάνεια. Θέλουν να προντήσουν περισσότερο την ασφάλεια και ίσως ξέρετε ότι τον Αύγουστο το Ισλαμικό κράτος μπήκε στον Βόρειο Λίμανο σε κάποια πόλη. Εκεί που είχαμε 45.000 καταγεγραμμένους πρόσφυγες. Πολύ αποστεθεροποιητικό αυτό για τη χώρα. Οπότε, είπαμε τώρα, χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια σε δήμους και κοινότητες για να περιορίσουν τους ε, πρόσφυγες και γι' αυτό και τώρα ζητούν περισσότερη βοήθεια από την διεθνή κοινότητα διμερή υποστήριξη. Τελευταίους μήνες, επίσης, διαπιστώσαμε ότι τώρα έχουμε κάποιους περιορισμούς εισόδου στη χώρα, Οπότε και ο αριθμός των προσφύγων που πήγαν στη χώρα τώρα έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Και οι πινακίδες ε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ που τους ε, χορηγούσαν. Κάτουν τώρα ένα μήνα. Τέλος πάντων δεν έχουμε αύξηση των προσφύγων. Οπότε τώρα διασκεδάστηκαν ε, οι φόβοι και ανησυχίε της χώρας. Αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα 100% γιατί ακόμα κάποιοι θέλουν οι πρόσφυγες να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Και ξέρετε βέβαια ότι στη Συρία κατάσταση μόνο σταθερή δεν είναι. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται για αυτούς που υποδέχθηκαν, τα κριτήρια υποδοχής που ε, δεν είναι σαφή και πώς θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για να υπάρχει κάποια στα σύνορα και δεν θέλει η κυβέρνηση πιο αυστηρή πολιτική όσον αφορά τα της ε, κατοικίας των προσφύγων. Ε, υπάρχει και θέμα με τα έγγραφα που έχουν ή δεν έχουν οι πρόσφυγες γιατί πρέπει να πληρώσουν κάποια τέλη που δεν έχουν τα πέρα τα χρήματα. Οπότε έχουμε αυτά τα προβλήματα. Για κοιτάξτε τώρα όλα αυτά πόσο αποσταθεροποιητικά είναι. Μια που οι πρόσφυγες αισθάνονται και αυτοί όλο ένα και περισσότεροι ανασφάλεια οι πρόσφυγες στο Λίβανο. Να, τι προβληματίζει τον κόσμο γιατί δεν θέλουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν αποξενωμένοι από τον τόπο που μένουν. Τώρα, κατά τα λοιπά για το Λίβανο, ίσως ενδιαφέρουν τα εξή. Ναι, μου φαίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η διαφάνεια. Είναι μια παραμεθορία περιοχή, εκεί που έχουμε κάποιους καταβλισμούς, που είπαμε πρόσφυγες μένουν παντού και έχουμε κάπου 70% των προσφύγων που ζουν σε τέτοια στρατόπεδα. Τα έχουν φτιαχτεί αυτά στο, στο γόνατο, δεν, δεν, δεν έχουν επίσημο χαρακτήρα. Και πολλοί από αυτούς τους κατακλυσμούς βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Βλέπετε κάποιοι από αυτού έπρεπε να φύγουν, τους πέταξαν έξω. Και μιλούμε για μία απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Εκεί όπου υπάρχει αντιπαράθεση, σύγκρουση. Γιατί πολλοί περνούν τα σύνορα και πάνε να μείνουν σε αυτά τα στρατόπεδα που είναι κοντά στα σύνορα. Οπότε, το θέμα είναι τι γίνεται εκτός αυτής της περιοχής. Ε, ας πούμε στα 10 χιλιόμετρα από τα ε, σύνορα. επομένω. δεν μπορούν παρά να νιώσουν ανασφάλεια οι Λιβανέζοι λόγω του πολέμου στη Συρία. Φοβούνται ότι ο πόλεμος πρόκειται να μεταδοθεί τώρα, να έρθει και στη χώρα τους. Όσον αφορά τώρα τις ανάγκες, δεν θα σας εκπλήξει να σας πω ότι οι περισσότεροι αυτούς που έφτασαν τελευταία χρονιά έχουν μετακινηθεί πάνω από μια φορά μέσα στην ίδια τους τη χώρα και επομένως για αυτούς είναι το τελευταίο καταφύγιο. Ο Λίβανος έχουν χάσει την οικογένεια, έχουν χάσει ό,τι είχαν στη ζωή τους, τα σπίτια τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι σημαδεμένοι για πάντα από αυτά που είδαν, από αυτά που υπέστησαν και έχουμε ας πούμε 30% των οικοκυριών που έχουν επικεφαλής γυναίκα. Πολύ δύσκολο αυτό για τις μητέρες αυτές που προσπαθούν να κάνουν τις ανάγκες των παιδιών τους χωρίς να έχουν σύζυγο. Οπότε ανασφάλεια και από εκεί. Το 39% των προσφύγων επίσης έχουν κάποιες ανάγκες συγκεκριμένες. Αυτοί που έχουν υποστεί κάποια αναπηρία μπορεί να είναι και ανήλικοι, τραυματίες, ε, έχουν βασανιστεί, έχουν υποστεί κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση. Φανταστείτε, ένα εκατομμύριο που δεν έχουν πρόσβαση ε, στις υπηρεσίες υγείας που είναι σχετικά υπηρεσίες ακριβές στον ε, Λίβανο. Οπότε ε, χρειάζεται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι έχουμε μπορέσει να τους καλύψουμε από αυτή τις υπηρεσίες υγείας και μιλάμε για 90.000 κάθε μήνα. Αλλά δεν μπορούμε να καλύψουν τίποτα παραπάνω από τα κατεπήγοντα περιστατικά, σωτηρία ζωής κλπ. Να έχουμε και εδώ ένα παιδί το οποίο έπεσε την σε όλο το σώμα λόγω μιας νάρκης, ενό όλμου που έσκασε στο σπίτι του, τον ε, σε μια ε, κουβέρτα γονεί, τον πήραν στο Λίβανο. Να, έγινε προσπάθεια ανακατασκευής του ε, προσώπου. Να, τι μας θυμίζει, γιατί χρειάζεται να μας θυμίζει το τι σημαίνει ο πόλεμος αυτός, πόσο τραυματικός είναι για την ανθρωπινή ζωή τώρα. Όσον αφορά τη διατροφική αρρωγή, έχουμε το 70% που έχουν βοήθεια σε αυτό το επίπεδο, από τη UNICEF, από την ε, Πάτη Αρμοστία κλπ. Οπότε χρειάζονται αυτή τη βοήθεια για τις βασικές διατροφικές ανάγκες και ε, έχουμε σχετικό διατροφικό πρόγραμμα αλλά έχει υποστεί το πρόγραμμα αυτό περικοπές. Αυτό το οποίο θέλουμε να υπάρξει είναι στρατηγικές και υπάρχει πίεση να πιάνουν να δουλέψουν οι ανήλικοι, να παντρεύονται οι μικροί κλπ. Το 31% που είναι πολύ, μιλάμε για το εκατομμύριο ζουν σε κάποιες κατοικίες που δεν έχουν καμία ασφαλή. Να βλέπετε εδώ μια φωτογραφία μια τέτοια σκηνής. Ε, οπότε έχουμε 17% που ζουν έτσι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει η κυβέρνηση, δεν επιτρέπει καταβλισμούς στρατόπεδα επίσημα για να μην τους ενθαρρύνουν να έρχονται και να μένουν και επομένως έχουν περιοριστεί προσπαθειές μας να τους δώσουμε ε, κουβέρτες, ε, ξύλα, τόσο κάτι για να μπορούν να ζεσταθούν αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την επιβίωσή τους αξιοπρεπή. 82% πληρώνουν κάποιο είδους νίκη, το οποίο είναι ένας τζίρος 43 εκατομμυρίων για το Λίβανο. Κάθε μήνα. Και αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται και κάποια κέρδη. Όλα αυτά πηγαίνουν στο λιβανισκό λαό. Αλλά από την άλλη μεριά φυσικά αυτό είναι πενταροδεκάρα σε σχέση με τη ζημία που έχουν υποστεί. Οπότε βλέπουμε πόσο σοκάρουν αυτά τα στατιστικά. Έχουμε δηλαδή 400.000 ε, παιδιά τα οποία είναι εκεί και είχαν πέρσι μόνο 300.000 τέτοια παιδιά ε, τα δημόσια γιατί όλοι οι υπόλοιποι θέλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως έχει σταθεί πάρα πολύ γενναιόδορη σαν εταίρος γιατί έχει βοηθήσει και μπορείς να βοηθήσει περίπου 100.000 παιδιά στα δημόσια σχολεία επειδή συμφώνησε το Υπουργείο Παιδείας. Πάντα είπαμε ε, με οικονομική επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το θέμα ότι ακόμα έχουμε 300.000 παιδιά που δεν έχει. Και επομένως αυτό είναι μια τραγωδία. Και αυτό δεν είναι θέμα ότι έγινε φέτος. Έγινε και πέρσι, έγινε και πρόπερσι. Αλλά έχουμε μία κούρση ενάντια στον χρόνο για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα έχουν κάποιο μέλλον αυτά τα παιδιά. Να μην είναι δηλαδή μία χαμένη γενιά. Οπότε... Μερικοί θα ενδιαφέρεστε για τη μετακατάσταση. Έχουμε ε, στόχο 130 ε, σύρους πρόσφυγες να ε, μετακατασταθούν μέχρι το 2016 και περίπου 100.000 είναι οι υποσχέσεις που έχουμε λάβει, όχι μόνο σε προγράμματα μετεκατάστασης, αλλά και ανθρωπιστικά προγράμματα ε, πανειστοχής, όπως ε, η Γερμανία για παράδειγμα, και πολιτικές ε, παραχώρησης θεωρήσεων. Είναι αυτονόητο ότι είναι πολύ σημαντικές τέτοιες πολιτικές και σημαντικά μηνύματα επιμερισμού του βάρους της ευθύνης σε περισσότερες χώρες, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους πρόσφυγες ε, να αισθανθούν ότι είναι πρόσδεκτοι και σε άλλες χώρες εκτός της, ε, της περιοχής. Και πριν ολοκληρώσω, να πω ότι σχεδιάσαμε τα προγράμματά μας προκειμένου να δρομολογούνται από δημόσιους φορείς και θεσμούς, ότι ό,τι γίνεται για τους πρόσφυγες να ωφελεί και τις λιβανέζικες κοινότητες. Και εδώ να τονίσω τον κρίσιμο και κέριο ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης και το δημιουργικό τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις ε, συνεισφορές που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χάρη σε αυτές ε, εξασφαλίσαμε στήριξη όχι μόνο για τα δημόσια σχολεία, αλλά και για τα νοσοκομεία, για κλινικές και τοπικά κέντρα. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε κάποια σχέδια στήριξης τοπικών κοινοτήτων ε, για εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές νερού, υπηρεσίες συγκομιδής απορριμμάτων σε κοινότητες που δεν είχαν τέτοιες υπηρεσίες. Και χάρη στους πρόσφυγες είχαμε βελτίωση της ζωής και της τοπικής κοινότητας. Έτσι κατευνάστηκαν κάπως οι εντάσεις εντός του Λιβάνου. Βέβαια οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι τεράστιες. Δεν λαμβάνουμε ε, τόση βοήθεια όσοι θα θέλαμε εξαιτία της πολιτικής ίσω κατάστασης, αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει τόσους πολλούς πρόσφυγες σε σχέση με το δικό της πληθυσμό. Είναι πολύ σοβαρέ αυτές οι αναλογίες. Επίσης, ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ενίσχυση, έχουμε και ανθρωπιστική ενίσχυση και αναπτυξιακή αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερη. Είναι κέρια σημασία ε, για το Λίβανο. Οι περισσότεροι πρόσφυγε ε, βρίσκονται σε περιοχέ ε, που το 68% των Λιβανέζων είναι φτωχοί. Αυτό δείχνει ο χάρτη. Και επίση συνεργαζόμαστε με 71 οργανισμού εντό του Λιβάνου και πρόσφατα απευθύναμε μία έκκληση για ένα σχέδιο ανταπόκρισης στο πρόβλημα των προσφύγων βλέπετε, και είναι δύσκολο βέβαια να ξεχωρίσετε από μακριά, βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει η χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική κρίση σε σχέση με πέρυσι, παρόλο που έχει διαπλασιαστεί ο προσφυγικός πληθυσμός. Και μάλιστα φέτος είναι κάπως αρνητικά τα πράγματα, χειρότερα από πέρυσι. Αυτά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, λέει αν θα ακούσουμε τώρα την κυρία Λόχπιλερ και τον κύριο Βάιτεν Χόλτσερ πρώτα και μετά να δώσω το λόγο στους για να υποβάλουν ε, ερωτήσεις. Οι κυρίες προηγούνται, λέει ο κύριος Βάιτεν Χόλτσερ. Κυρία Λόχπιλερ, οι κυρίες προηγούνται, όπως ακούσατε. Εμείς ε, περάσαμε τρεις ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα στην Βηρητό και στο Λίβανο. Σας ευχαριστούμε πολύ βεβαίως και εσάς του είπα του αρμοστή των ε, Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες που μας κάνατε την ενημέρωση. Είδαμε βεβαίως και τους, τον πρέσβη, μας βοηθήσατε βεβαίως και με την ε, διοικητική οργάνωση. Βεβαίως είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πήγαμε στην κοιλάδα Μπεκά που είναι βεβαίως ο στοβολώνας της περιοχής και εκεί είναι ορατό, πολύ ορατό. Οι Λιβανέζοι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη στρατόπεδα για να μην εξισωθούν με τους Παλαιστινίους πρόσφυγες που έμειναν εκεί για πάντα, έτσι χρησιμοποιούν άλλες λέξεις. Παρ' όλα αυτά οργάνωσαν, πώς να το πω, αυτά τα στρατόπεδα και λειτουργούν. Όμως το τοπίο και τα χωριά είναι γεμάτα καλυβούλες και άλλα πρόχειρα παραπήγματα Πώς ε, μπόρεσαν οι άνθρωποι να περάσουν τις τρεις αυτές βαριές κακοκαιρίες του φετινού χειμώνα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα εξηγήσατε ήδη. Νομίζω ότι η λιβανική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Λιβάνου αξίζει ευχαριστίες διότι επέτρεψε την είσοδο των ε, προσφύγων. Ένας από τους τέσσερις σημερινούς κατοίκους του Λιβάνου είναι πρόσφυξη. Πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια. Τώρα βέβαια Υπάρχουν και συστάσεις προς ε, τις λιβανικές αρχές και τον UNHCR να κάνουν κάποιες αλλαγές. Αν έχετε, αν είσαστε καταχωρισμένος πρόσφυγας, οφείλετε μετά να υποσχεθείτε, ε, να δώσετε το λόγο σας δεν θα εργαστείτε. Βέβαια, οι ανάγκες που έχουν είναι βασικές. Και κάθε έξι μήνες το κάθε νοικοκυριό πληρώνει 200 δολάρια κάθε έξι μήνες. Ε, πού θα βρείτε τα χρήματα ως πρόσφυγας δηλαδή για να διατηρήσετε την ιδιότητα του πρόσφυγα αφού πρέπει για να καταχωριστείτε ξανά κάθε πρόσωπο πάνω των 15 ετών της οικογένειας να πληρώνει 200 ευρώ όπως είπα περίπου. Υπάρχει τώρα και αυτό, αυτή η ρύθμιση για τα σύνορα για τους ε, σύρους πρόσφυγες από το Γενάρη νομίζω. Βεβαίως λειτουργούν καλύτερα οι μεθοριακοί έλεγχοι όμως αυτό σημαίνει καμιά, βαριά, καμιά φορά βαρύτατες καταστάσεις. Οι πρόσφυγες από τη Συρία έχουν μάθει ότι το κράτος οργανώνει την υγεία, η οποία είναι δωρεάν. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει στο Λίβανο. Μία οικογένεια με πέντε παιδιά. Ένας από τους γονιούς έπαθε καρκίνο. Δεν έχουν χρήματα λοιπόν για να πληρώσουν τη θεραπεία στο Λίβανο, αναγκάζονται να περάσουν τα σύνορα, αφήνουν τα παιδιά πίσω για να ε, ε, πάνε για να κάνουν θεραπεία στην Συρία. Δεν του επιστρέπουν να επιστρέψουν στο Λίβανο μετά. Και σε άλλη υπόθεση μπήκε και στις εφημερίδες εκεί κάποιες συριακές κοινότητες που καταλήφθηκαν από μαχητές του Ισλαμικού κράτους όμως οι αρχές ε, του Λιβάνου κάνουν στραβά και τους βοηθούν για να έλθουν έτσι λοιπόν οι Συριακές οικογένειες βρήκαν που να μείνουν τελικά. Κάποιοι από τους ακτιβιστές, ας το πω έτσι, μας είπαν ότι πρέπει να φτιαχτεί μια πολιτική για τους Σύρους πρόσφυγες, γιατί αυτοί είναι ακόμα σε κομμάτια. Και ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ να βοηθήσει. Επίσης, ο UNHCR μπορεί να κάνει περισσότερα να εκπαιδεύσει τον κόσμο για το δίκαιο των προσφύγων, πρόσωπα δηλαδή που εργάζονται σε μεθοριακά γραφεία, καθώς επίσης και σε τοπικές κοινότητες, διότι κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά. Για μας τώρα τις χώρες μέλη της Ένωσης, είπατε και εσείς ότι 39% των ε, προσφύγων έχουν ειδικέ ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες μέλη να προωθήσουν αυτό το πρόγραμμα επανεγκατάστασης που έχετε φτιάξει και που λαμβάνετε κάποια χρηματοδότηση από την Ένωση και που μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Και όπως είπατε επίσης, βέβαια, υπάρχει ανταγωνισμός των προσφύγων με τους ντόπιου. Και οι Σύριοι είναι θαυμάσιοι επιχειρηματίες. Αυτοί οι μικρομεσαίοι που φτιάχνουν μια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό και δεν υπάρχουν ρυθμίσει για τον ανταγωνισμό αυτό και επίση τα επίπεδα του πολύ χαμηλού εισοδήματο, και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός με του κατοίκου τη υπαίθρου. Αυτό εντείνει τι εντάσει αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται μια γενικότερη πολιτική προσέγγιση. Το πρόγραμμα της παιδείας, επίσης, τελικώς θα υπάρξει μια χαμένη γενιά. Ο UNHCR υπολόγισε ότι χρειάζονται 650 δολάρια για κάθε παιδί το χρόνο για να πάνε στο σχολείο. Όμως φέτος μόνο 60.000 Σύριοι πρόσφυγες, πάνε ε, στα σχολεία με στόχο να γίνουν 150.000. Όμως αν δεν υπάρχει σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης γιατί όσοι οι Σύριοι πρόσφυγες έχουν περισσότερα χρήματα στέλνουν τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πρόβλημα παιδείας γιατί θα είναι όπως είπα μια χαμένη γενιά και βεβαίως αυτή θα είναι ανοιχτή σε ε, φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης. Μου επιτρέπετε τώρα να περάσω το λόγο στον ε, συνάδελφό μου. Μια στιγμή λέει πρόεδρος. Γιατί έχουμε επισκέπτες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επισκέπτες. Αλλά παρακαλώ καθίστε, μη και στα όρθιοι. Χαίρομαι που ήρθατε. Βλέπετε ότι υπάρχουν καινέ θέσει. Καθίστε. Por favor, siéntense porque es difícil hablar. Μη καθίστε. Gracias. Κύριε Χόλσερ συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Λοχπίλερ. Όλοι εντυπωσιαστήκαμε από τα όσα συμβαίνουν στο Λίβανο και ιδίως ότι ο λιβανικός λαός έχει αναλάβει τρομερές επιβαρύνσεις. Ένα τέταρτο μέχρι σχεδόν το ένα τρίτο του κόσμου που διαμένει αυτή τη στιγμή στο Λίβανο είναι πρόσφυγε πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται όμως απόλυτα ξεκάθαρα νούμερα διότι την καταχώρηση, την καταγραφή την κάνει ο UNHCR και μετά αυτά τα δεδομένα μετα... διαβιβάζονται στην κυβέρνηση και ίσως γίνονται, παραβλέπονται κάποια πράγματα. Διαπιστώσαμε επίσης κάτι που είναι ανησυχητικό, ιδίω σε συζητήσεις με πρόσωπα που βρούν στον χώρο των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και δικηγόρους, ότι οι εντάσεις ανάμεσα στα τμήματα του πληθυσμού, δηλαδή των Λιβανέζων και των προσφύγων, ότι οι εντάσεις αυτές μεγαλώνουν. Είναι θέμα βεβαίως και dumping αμοιβών και μισθών. Είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι έρχονται και εργάζονται πλέον υπό απίστευτες συνθήκες έχουν όμως ανάγκη από τα λεφτά, οπότε κάνουν, αναλαμβάνουν δουλειές που τους φέρνουν τελικά σε αντίθεση με τον τόπιο πληθυσμό, το ίδιο και με καταστήματα. Κατηγορούν επίσης τους πρόσφυγες ότι αυτοί φταίνε που υπάρχουν διακοπές ρεύματος στο Λίβανο. Τους κατηγορούν επίσης ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα. Όλα αυτά δεν φαίνεται να είναι αλήθεια. Όμως είναι εντάσει που οφείλει να καλάβει κανεί σοβαρά υπόψη. Τα δείξατε κι εσείς πόσο γρήγορα μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα αυτά. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να αντέξουν οι άνθρωποι αυτή την κατάσταση. Εγώ αμφιβάλλω αν μπορούν να αντέξουν έστω και ένα χρόνο παραπάνω. Υπάρχουν και αυτοί οι μεθοριακοί έλεγχοι, όπου οι συνομιλητές μας μας είπαν ότι οι άνθρωποι που διαβαίνουν τα σύνορα τώρα έχουν περιοριστεί διότι δεν είναι πλέον τόσο έντονες οι συγκρούσεις στη Συρία ώστε να προκαλούν σημαντικά ρεύματα προσφύγων προς την πλευρά του Λιβάνου. Όμως υπονοούν ταυτόχρονα ότι αν ενταθούν πάλι συγκρούσεις αυτές θα δυναμώσουν πάλι τα ρεύματα αυτά. Και το ερώτημα πάντοτε που τέθηκε στις συζητήσεις αυτές είναι με το πιο ενδιαφέρον και συμφέρον έχει η λιβανική κυβέρνηση η κατάσταση αυτή να παραμείνει προσωρινή και όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς να φύγουν να πάνε στην Ευρώπη. Μιλήσαμε και με τους σύρους χριστιανούς οι οποίοι λένε με μεγάλη ανησυχία ότι δεν θέλουν να φύγουν ακόμα περισσότεροι σύροι χριστιανοί και να μεταβούν στο Λίβανο. Το ερώτημα εν τέλει είναι τι μπορεί να κάνει κανείς και γιατί αριθμούς πρέπει να μιλεί κανείς εάν θέλει να συζητήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Και τέλος, το θέμα της χρηματοδότησης. Βεβαίω η Ευρώπη, είπατε και εσείς, κάνει πολλά πράγματα. Αν όμως το πρόγραμμα ΕΚΟ δίνει 23 εκατομμύρια ευρώ, αλλά βεβαίω λέτε και εσείς ότι αυτά τα ποσά πόρο απέχουν από το να εξασφαλίζουν τους πόρους που έχει ανάγκη ο UNHCR. Ωστόσο θα ήταν καλή επένδυση από πλευρά της Ευρώπης να κάνει περισσότερα πράγματα. Η ΔΕΜΗ πώς θα αντέξει την πίεση αυτή και ποιος θα την αντέξει. Ίσως είναι πολύ βραχυπρόθεσμη η μνήμη μας. Αλλά μην δυσμονούμε ότι ο Λίβανος πέρασε από ένα 15 ετή εμφύλιο πόλεμο και αυτός δεν έχει τελειώσει και τόσο πολλά χρόνια. Υπάρχουν και τα στρατόπεδα των Παλαιστινίων. Πολλοί μας είπαν ότι τώρα ίσως να συμβεί ξανά το ίδιο και ότι λίγο πολύ μπορεί να καταλήξει η κατάσταση αυτή πάλι σε εμφύλιο πόλεμο στον Λίβανο εάν πάρουν στραβό δρόμο οι εξελίξεις. Έτσι λοιπόν, ναι μεν είναι μεγαλειώδες αυτό που πετυχαίνει η διεθνής κοινότητα, αλλά φοβούμαι ότι χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους πόρους και εμείς και ως ευρωβουλευτές έχουμε και το καθήκον και την υποχρέωση να τα πούμε τα πράγματα αυτά. Αλλιώς εκεί κάνει τικ-τακ μια ορολογιακή βόμβα η οποία μπορεί κάποτε να εκραγεί και να κάνει μεγάλη ζημιά και στην Ευρώπη, αν δεν δράσουμε ήδη από τώρα. Ευχαριστώ. Ποιος συνάδελφος θέλει το λόγο παρακαλώ. Μέχρι τις 5 και 4 θα δίνω το λόγο στους συναδέλφους και κατόπιν στην κυρία Κέλλη για να απαντήσει. Η κυρία Βίμπερκ, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για το καταπληκτικό έργο που επιτελεί και θα πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την Υπα-Τιαρμοστία γιατί και αυτή η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών υποφέρει και με ελάχιστα χρήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και είναι τεράστια η ευθύνη που έχει αναλάβει ο Λίβανος, υπερβολική και ακούσαμε από τους προλαλήσαντες ότι άρχισε και δημιουργούνται κάποιες εντάσεις. Άκουσα για μια οικογένεια που ο πατέρας ήταν οικοδόμος και τώρα έχει χάσει τη δουλειά του γιατί ένας πρόσφυγας ε, κάνει την ίδια δουλειά με πολύ λιγότερη αμοιβή. Οπότε χάνει το εισόδημα, το βιοπορισμό του η οικογένεια αυτή και βλέπουμε ότι και ο τοπικός πληθυσμός μερικές φορές υποφέρει από αυτή την αθρώαση ροή των προσφύγων. Θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα αναλάβουμε και εμείς ευθύνες μας, γιατί είναι δύσκολο όταν ο ίδιος ο πληθυσμός ο Λιβανικός υποφέρει να αφιερώνει ταυτόχρονα η χώρα αυτή χρήματα για τους πρόσφυγες να τροφοδοτεί την ύπατη αρμοστία. Τι περιμένει λοιπόν η ύπατη αρμοστία από εμά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε περισσότερα κονδύλια, θέλετε να υποδεχθούμε περισσότερου πρόσφυγε εμεί στι δικέ μα χώρε. Είπαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου. Και πρεσβείε σε διάφορε χώρε για να μπορεί κανεί να ζητά ανθρωπιστική βίζα. Είναι ε, δική σα μια τέτοια έκκληση, πιστεύετε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. E, και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την εισήγησή σας. Μας βοηθά να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας αλλά και να βελτιώσουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε. Πάντως, θέλω να σας πω ότι είμαι συνεισηγήτρια για τη στρατηγική έκθεση της πρωτοβουλίας όσον την κατάσταση στην Μεσόγειο και την ανάγκη μιας σφαιρικής προσέγγισης της ε, Ένωσης όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, θα καλύψουμε πάρα πολλά θέματα, ε, την επανεγκατάσταση και άλλα θέματα όπως την έρευνα και διάσωση, την εφαρμογή του άρθρου 80 και άλλα θέματα που αφορούν το εσωτερικό και το εξωτερικό ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει συνεργασία τις αμέσως επόμενες εβδομάδες είπατε και πέστε μας εσείς τι προς το κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ούτως ώστε να έχετε κάποια πολύ συγκεκριμένη ανταπόκριση πέραν της έκθεσης αλλά συγκεκριμένα πώς πέστε μας συγκεκριμένα σε ποια σημεία μπορούμε να προσπαθήσουμε και να πώς να το λύσουμε τις επιλογές μας. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλη. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την παρουσίασή σας και να σας διαβεβαιώσω για το τεράστιο σεβασμό που τρέφουμε προς την οργάνωσή σας στην υπακερμοστία. Και επίσης ε, τρέφουμε ιδιαίτερο θαυμασμό και σεβασμό προς τη λιβανική κυβέρνηση. Και μάλιστα η σύγκριση που κάνατε με το Βέλγιο με συγκλώνησε, γιατί και εγώ Βέλγος είμαι. Και μπορώ να φανταστώ ότι τεράστια πίεση ασκείται στην τοπική κοινωνία από την αθρώα αυτή προσέλευση των προσφύγων. Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες έχουν σειρεύσει στο Λίβανο, σε μια τόσο μικρή χώρα. Και είπατε ότι ήταν αρκετά τεραχώδες και το παρελθόν στη χώρα αυτή. Οπότε ερωτώ, σε ποιο βαθμό αυτή η μαζική προσέλευση προσφύγων στο Λίβανο έχει αλλάξει την πολιτική και την θρησκευτική κατάσταση στη χώρα. Γιατί είναι δύσκολη ανέβριση ισορροπιών εκεί και ίσως είναι εύκολο να δημιουργηθεί ανισορροπία. Πώς επηρεάζει λοιπόν την γενικότερη πολιτική και κοινωνική κατάσταση στο Λίβανο η έλευση των προσφύγων. Εμείς βέβαια και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας ε, συνεισφέρουμε ε, στην περιοχή και στηρίζουμε την υπατηρμοστία. Αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα τώρα, ε, ποια είναι η πιο κατεπίγουσα και επιτακτική ανάγκη, οικονομική, χρειάζεται κονδύλια ή θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα παράλληλα. Και πώς ε, κρίνετε τις διεθνείς προσπάθειες και την πρόταση για υποδοχή σύρων προσφύγων και από άλλες χώρες. Είναι αρκετές οι χώρες που είναι διατεθειμένες να ανοίξουν τα σύνορά τους προς τους σύρους ή αυτό που προέχει είναι να βρεθούν πόροι και κονδύλια ώστε όπου και αν βρίσκονται οι σύροι πρόσφυγες να βοηθούν οι χώρες για να τους προσφέρουν προστασία. Βέβαια, το καλύτερο σενάριο θα ήταν ε, να τεθεί ένα τέρμα στην έναπλη σύραξη της Συρίας και να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες προοπτικές ώστε να μπορέσουν να επαναπατριστούν όλοι αυτοί οι Σύριοι πρόσφυγες. Βέβαια αυτό προς το παρόν είναι ένα όνειρο. Και βραχυπρόθεσμα μάλλον απατηλό. Γιατί Δυστυχώς συνεχίζεται η ένοπλη σύραξη, οπότε συνεχίζεται η μεταναστευτική πίεση και διερωτόμαστε πόσο θα αντέξουν οι γειτονικέ χώρες, πόσο καιρό θα μπορούν να δέχονται και να απορροφούν αυτές, αυτά τα κύματα προσφύγων. Γιατί είπατε ότι ουσιαστικά ο Λίβανος έκλεισε τα σύνορά του. Ενώ οι Σύριοι εξακολουθούν να θέλουν να γλιτώσουν από τη χώρα για να σώσουν τη ζωή τους. Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η προοπτική. Μια στιγμή κυρία Κέλλη. Έχουμε και τον ε, πρώτο γραμματέα της ε, πρεσβείας του Λιβάνου στη συνεδρίαση. Θα σας δώσω το λόγο για τρία μόνο λεπτά δυστυχώ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλώς ορίσατε και παρακαλώ έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ κυρία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποια θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την σημερινή συνάντηση. Πρώτα πρώτα, να σας πω τι γίνεται με αυτό το έγγραφο πολιτικής της κυβέρνησης που ανάγεται στο 2014 και θέλω να σας τονίσω ότι αυτό το έγγραφο μιλάει για εξασφάλιση της ασφάλειας και συρρήγνωση των αριθμών, συρρήγνωση των μεταναστευτικών ροών. Έχουμε κάποια εμπειρία σχετικά με αυτά και νομίζω ότι και η κυρία Κέλλη γνωρίζει την εμπειρία μας. Οπότε τώρα υπάρχουν ε, προσδοκίες σε σχέση με τους ε, πρόσφυγες. Ελπίζει ο κόσμος ότι θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Ε, ενώ είναι γνωστή η κατάσταση στη Συρία. Πάντως η θέση μας είναι να δούμε τις τρεις βιώσιμες λύσεις όταν έρθει η ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως προς το παρόν κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να παράσχουμε διεθνή προστασία. Παρά το ότι δεν έχουμε προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1951 περί προσφύγων. Όσον αφορά την ε, ανανέωση της άδειας ε, διαμονής πρόκειται για τυπικές διαδικασίες για τους πρόσφυγες ή για τους ετούντες άσυλο και πάντα χρειάζεται να υποβάλλονται κάποια έγγραφα. Όταν δεν έχει ο ετών ε, έγγραφα θα πρέπει να έχει κάποιο άλλο επίσημο αποδεικτικό. Πάντως, εγώ θα πρέπει να σας τονίσω ότι ο Λίβανος έχει ένα σχέδιο αντιμετώπιση τη κρίση. Το έχει υπόψη τη είπα διαρμοστή, μπορεί η κυρία Κέλλα να μας πει δύο λόγια για αυτό. Τρόσον να αφορά το καθεστώ που τους διέπει και το πώ θα πρέπει αυτό να περιχαρακωθεί, να ξεκαθαριστεί. Ξέρουμε ότι κάνει πάρα πολλά σχέδια με αυτό η πατιαρμοστία και την ευχαριστούμε. Πάντω, Συνήθω είναι αρμοδιότητα του κράτου να προωθήσει, να περιώσει τις αιτήσει των όσων ψάχνουν άσυλο. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ που λάβατε το λόγο και που ήρθατε κι εσείς να βάλετε το λιθαράκι σας. Κυρία Κέλλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Λιβάνου, τον οποίο συγχαίρω επίσης για τα εκπληκτικά επιτεύγματα της κυβέρνησης της χώρας σας. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανος. Εγώ μάλιστα θεωρώ ότι είναι προνόμιο για τον εαυτό μου που μπορώ και εργάζομαι εκεί και τα βλέπω ίδια. Θα έρθω τώρα σε, ορισμένα, σε ορισμένες μάλλον από τις παρεμβάσεις με τη σειρά που τις άκουσα. Όσον αφορά την εκπαίδευση ε, προσωπικού στα σύνορα και στις τοπικές κοινότητες. Προχωρούμε, έχουμε και σχέδιο μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών για να φτιάξουμε τη λεγόμενη capacity building και με τους τοπικούς αστυνομικούς και στις κοινότητες, τοπικές κοινότητες. Βοηθεί εκεί το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και η δύναμη εσωτερικής ασφάλειας. Και είναι μάλιστα και ένα project το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι εδώ. Επίσης συζητούμε και συνεργαζόμαστε και με το Υπουργείο κοινωνικής πρόνοιας για την διευκόλυνση των προσώπων που διαβαίνουν τα σύνορα. Επίσης, η δημόσια παιδεία. Έχουμε ήδη 100.000 παιδιά στα δημόσια σχολεία και μάλιστα έχει αυξηθεί ο αριθμό αυτό τι τελευταίε εβδομάδε. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδεία πάλι σε πολύ επικοδομητική προσπάθεια, τη οποία ηγείται ο ίδιο ο Υπουργό, συγκεντρώνει δωρητέ και από τον Οργανισμό ε, Ενωμένων Εθνών και τοπικούς παράγοντες με στόχο να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μέσω της παιδείας και να φτάσουμε στο το 2016 σε 400.000 παιδιά στα σχολεία. Βέβαια το κόστος παιδί που το έχει δεχθεί και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι σχετικά υψηλό. Είναι περίπου 600 δολάρια το κάθε παιδί στη δεύτερη βάρδια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πόρους. Χρειάζονται πόροι. Αυτό όμω είναι και ο στόχο. Στήριξη των δημόσιων θεσμών για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Έχουμε και 300.000 παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ επιλογέ και για αυτά. Πάλι εκεί, μέσω του Υπουργείου Παιδεία, προχωρούμε και κάποιε non-formal options. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα, είναι αληθέ ότι ο ύπατο αρμοστή χρησιμοποιεί βιομετρική τεχνολογία για να καταχωρίζει και να καταγράφει όλου του πρόσφυγε. Επίσης επαληθεύουμε τους ε, ε, πρόσφυγες όταν εκπνέουν τα πιστοποιητικά τους. Τους φέρνουμε δηλαδή στις υπηρεσίες μας και, τους, ε, και επαληθεύουμε τα πιστοποιητικά τους πριν να τα επανεκδώσουμε. Αυτά τα κάνουμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε ο Λίβαρος να γνωρίζει ανά πάση στιγμή ποια πρόσωπα βρίσκονται στην επικράτειά του και το κράτος αναλαμβάνει και μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ε, ανταπόκρισης των πρόβλημα των προσφύγων. Και βέβαια υπάρχουν ε, εντάσεις, εντάσεις. Και βέβαια οι Σύριοι εκτοπίζουν το λιβανέζικο εργατικό δυναμικό κυρίως σε ε, θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων. Και βέβαια οι Σύριοι είναι τόσο απεγνωσμένοι που δουλεύουν σχεδόν τζάμπα και βεβαίως οι περισσότερες δουλειές που βρίσκουν είναι στον άτυπο τομέα και όπου δεν συγκεντρώνονται πολλοί Λιβανέζοι, για παράδειγμα στα γεωργικά και στις οικοδομές. Και άλλωστε όχι μόνο εμείς αλλά και άλλοι οργανισμοί λέμε ότι οι Σύριοι θα πρέπει να απαιτείται να σέβονται τους νόμους του Λιβάνου και Συνεργαζόμαστε επίσης με τους εταίρους μας και βρισκόμαστε σε συζήτηση και με κυβερνητικές υπηρεσίες για να δούμε τι είδους πολιτική εργασίας μπορούμε να εφαρμόσουμε για να προχωρήσει ο Λίβανος, να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στον Λίβανο και οι πρόσφυγες τελικά αντί να είναι τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη να συμβάλλουν σε αυτήν. Βεβαίως δεν είναι και εύκολο να το περάσουμε αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει ανταγωνισμός από πλευρά των προσφύγων για τις λίγες δουλειές. Πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη ευαισθησία. Όσον αφορά το τι θα συμβεί εάν υπάρξει και πάλι μαζική σώρευση προσφύγων, έχουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε μια αύξηση των προσφύγων, αλλά βέβαια μεγάλη, έντονη ε, προσέλευση προσφύγων θα είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο με φαίνει σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Η λύση για το πρόβλημα πρέπει να βρεθεί μέσα στην ίδια τη Συρία. Ένα από τα προβλήματα που δίνουν και το πρόσωπο στην τραγωδία που είναι ζωντανή μέσα στο μυαλό του καθενός είναι ότι μέχρι να υπάρξει λύση εντός της Συρίας θα χαθούν ακόμα αναρρύθμιτες ζωές. Οι άνθρωποι θα φεύγουν προς γειτονικέ χώρες. Οι γειτονικέ χώρες θα αποσταθεροποιούνται από τη σύγκρουση αυτή και τελικώς δεν φταίνε. Όσον, αφορών, όσον αφορά τώρα την οικονομική στήριξη, έχουμε, είναι αλήθεια, στήριξη από πολλά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ότι θα συνεχίσουν τη χρηματοδότηση αυτή. Λέμε σε όλες τις δωρήτριες χώρες και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η ανθρωπιστική χρηματοδότηση πρέπει να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Ο Λίβανος είναι χώρα μεσαίου εισοδήματο. Ε, τα δάνεια που έχει λάβει τώρα την αποκλείουν από το να λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση. Πάλι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει χρηματοδοτική υποστήριξη ανάπτυξη για πολλά χρόνια με πολλού και επικοδομητικού τρόπου. Έχει κρίσιμη σημασία αυτό να συνεχιστεί. Θα έλεγα λοιπόν, μάλλον με ρωτήσατε, τι προτεραιότητα να βάλω σε αυτά που θα ήθελα να κάνετε. Πρώτα, η πολιτική επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία. Αυτό θα πρέπει να είναι και το πρώτο, διότι αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να βάζουμε ένα τσιρότο πάνω σε μια πληγή που αιμορραγεί. Το ίδιο για το ανθρωπιστικό. Χωρίς την ανθρωπιστική υποστήριξη οι άνθρωποι θα πεθαίνουν σε μεγάλους αριθμούς. Και μόνο λόγω της ανθρωπιστικής στήριξης που έχουμε λάβει, χάρη σε αυτήν δηλαδή, μπορέσαμε να επιτύχουμε όσα επιτύχαμε. Και οι άνθρωποι να μην έχουν πληγεί ακόμα χειρότερα. Στήριξη για την ανάπτυξη. Στήριξη πως θεσμούς του Λιβάνου, αλλά και στο επίπεδο των κοινοτήτων. Υπάρχουν project με χαμηλή ανάγκη χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, ηλεκτρικές γεννήτριες, ε, αντλίες για το νερό, για την άρδευση. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν πολύ, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μείωση των εντάσεων στις τοπικές κοινότητες του Λιβάνου, γιατί μπορούν τότε οι Λιβανέζοι να δουν ότι δεν τους ζητούμε απλά να κάνουν περισσότερα, αλλά ότι έρχονται οι εταίροι τους και τους υποστηρίζουν, τους βοηθούν, τους προσφέρουν υπηρεσίες και μάλιστα που ορισμένες τοπικές κοινότητες δεν είχαν καν πριν από την ανθρωπιστική κρίση. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση, εδώ λέμε διάφορα πράγματα. Θα θέλαμε να δούμε οι θέσεις για επανεκατάσταση στην Ευρώπη να αυξηθούν σε αριθμό. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα αυτό. Το Humanitarian Admissions Program έχει πραγματικά δημιουργικό χαρακτήρα. Η αριθμή που δέχθηκε η Σουηδία έχει μειώσει τις απαιτήσεις, έχει χαλαρώσει τις απαιτήσεις για προξενικές θεωρήσεις, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες σε πρόσφυγες να έλθουν να ε, σπουδάσουν επίσης για θεραπεία στο άσυλο όπου Σύριοι πρόσφυγες φτάνουν στη χώρα και αντιμετωπίζονται με δίκαιο και ανθρωπιστικό τρόπο. Αυτά είναι κρίσιμη σημασία. Για την Μεσόγειο, ο UNHCR έχει συγκεκριμένες συστάσεις που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας, βεβαίως και με τους συναδέλφους μου εδώ στο γραφείο μας των Βρυξελών. Πολύ ευχαρίστως να συμμετάσχουμε σε ένα ρωμαλαίο διάλογο μαζί σας, να δούμε δηλαδή τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει ο δικός μας οργανισμός στο δικό σας προβληματισμό. Τώρα, πώς άλλαξαν την πολιτική κατάσταση στον Λίβανο οι ελεύσεις των προσφύγων. Εδώ μπορώ να πω ότι η κρίση της Συρίας έχει φέρει κοντά τους πολιτικούς ηγέτες με πολύ θετικό τρόπο. Είδαμε και πολύ συνένεση για το σχέδιο ασφάλειας, για τη σταθεροποίηση του Λιβάνου. Βεβαίως και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ τους, αλλά μέχρι τώρα αντέχουν οι άνθρωποι. Και αυτό οφείλεται σε αυτή την ενωτική προσπάθεια των Λιβανέζων. Πολλοί λένε ότι οι Λιβανέζοι είναι τους πιο ανθεκτικούς ανθρώπους στον κόσμο. Ο Λίβανος ως χώρα πέρασε από 15 ετή εμφύλιο πόλεμο και άντεξε. Και ακόμα είναι στη φάση της ανοικοδόμησης. Είναι άνθρωποι με γερή βιομηχανία, είναι άνθρωποι, συγγνώμη, μάλλον επιμελείς και ε, δουλευταράδες. Υπάρχει και το σχέδιο ανοικοδόμησης στο σχέδιο για την περιφερειακή αντιμετώπιση με παραπάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η διάσκεψη του Κουβέιτ που θα γίνει τούτο το μήνα είναι επίση πολύ σημαντική. Πέρσι 90% των υποσχέσεων από δωρητέ που έγιναν στο Κουβέιτ τελικώ στηρίθηκαν. Και αυτό μα επέτρεψε να έχουμε τη ροή αυτή τη χρηματοδότηση. Και αυτό έχει και συμβολικό χαρακτήρα τώρα. Γνωρίζω ότι έχουν εγκριθεί πολλέ από τι δαπάνε αυτέ, αλλά μην λησμονείτε τη μικρή αυτή περιοχή του κόσμου που έχει επομιστεί ένα δυσανάλογο βάρος της οποίας όμως αυτής της περιοχής του κόσμου η σταθερότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ πέραν της περιοχής όπου βρίσκεται. Και βεβαίως θα έχει επιπτώσεις και στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν ελπίζω να απαντούν στις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να προσέλθω να συζητήσουμε για την ε, υπόθεση αυτή η οποία πραγματικά με απασχολεί βαθύτατα και νομίζω ότι όπως είπε και ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως του Λιβάνου, ο Λίβανος είναι μια σπουδαία, ένα σπουδαίο παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει με το πιο θετικό ανθρώπινο πνεύμα. Αλλά χρειάζεται και περισσότερη υποστήριξη σε μια τέτοια μικρή χώρα η οποία όπως είπα επομίζεται κάτι που είναι αδιανόητο για τους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Θερμές ευχαριστίες ε, για το τιτάνιο έργο σας και για το ότι είχατε την καλοσύνη να έρθετε και να μας το παρουσιάσετε. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας ε, στηρίζουμε όλη της ύλη. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλη. Σε levanta la sesión. Λύεται η ναι. συνεδρίαση.